So, ladies and gentlemen. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζω σε αυτή την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Δεύε. Χαιρόμαστε που έχουμε εδώ την κυρία Λίντα Μακάβεν, σας καλωσορίζουμε λοιπόν συνάδελφοι και εδώ συνήθω αυτή την αίθουσα κάνουμε τη συνεδριάση. Είμαστε στη θέμα 34 της ημερήσιας διάταξης και ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε στις 6.30 να τη συνεδρίαση γιατί κάποιοι από εμάς είναι εδώ από τις 9 το πρωί. Το πρώτο θέμα της κυρίας μας συνεδρίασης ε, αφορά τη μεριστή διάταξη. Αν δεν έχετε αντιρρήσει εγκρίνεται, δεν έχω ανακοινώσει και φτάνουμε στο 3 τώρα. Γιατί συνεδριάζουμε σήμερα, διότι θέλουμε να εξετάσουμε τις ε, τροπολογίες που αφορούν το μηχανισμό γειτονίας ανάπτυξης και διεθνούς Συνεργασίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα καθορίσει πώς η αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες της τάξης περίπου των 90 δις θα δαπανηθεί 21 με 27. Όπως ξέρετε, αυτή η κοινή συνεδρία γίνεται βάσει της διαδικασίας του άρθρου 55. Έχουμε τέσσερις συνσυντονιστές. Τον Κριστιαν Βαν τον Πιερ Παντζέριου, τον Φρανκ Έιντζελ και τον Σαρλ Γκρέμς. Έχουμε 997 τροπολογίες που πήραμε, εκτός από τις 380 που έχουν καταθέσει οι συνεισηγητές. Επίσης πρέπει να πω ότι έξι επιτροπές γνωμοδετούν για την έκθεση αυτή, συμπεριλαμβανομένη του Επιτροπής Προϋπολογισμού βάσει του άρθρου 54 και των γυναικών βάσει του άρθρου 53. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας και αποφάσισα οι συγκητές εξαιτίας αυτού του φόρτου εργασίας να αναβάλουν την ψηφοφορία από τις 4 Φεβρουαρίου στις 4 Μαρτίου, ώστε να μπορέσει να υπάρξει αρκετός χρόνος για να κατατεθούν συμβαστικές τροπολογίες. Επίσης ξέρουμε ότι ο μηχανισμός γειτονίας ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας και ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας είναι δύο μηχανισμοί οι οποίοι θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και δεδομένου ότι η ψηφοφορία του Μηχανισμού Προταξής βοήθεια θα γίνει στι 4 Φεβρουαρίου, η ευθυγράμμιση θα πρέπει να γίνει στι τροπολογίε που θα παρουσιαστούν στην Ολομέλεια. Δίνω το λόγο συνάδελφο. Σα ευχαριστώ. Πρέπει να σα πω ότι συναντήσαμε την Προεδρία τη Ρουμανική σήμερα και για το Ινδίκη μάθαμε τι ακριβώ σημαίνει στο Συμβούλιο. Τώρα, εάν θα πρέπει το EDF να συμπληρωθεί στον προπολογισμό ή θα πρέπει ε, να τα βάλουν όλα αυτά σε αυτό το οποίο λένε Nego Box, δηλαδή ένα κουτί διαπραγμάτευση, όχι σε Lego, δηλαδή κάποια σημαντικά θέματα τα αφήνουν να περιμένουν σε αυτό το κουτί μέχρι τον Σεπτέμβριο και ασχολούνται με άλλα θέματα πιο δευτερεύοντα ίσω. Ήταν λοιπόν σημαντικό να σα το πω αυτό. Αν θέλουμε εμεί η πρώτη ανάγνωση να ολοκληρωθεί πριν από τι εκλογέ, να ε, προχωρήσουμε ώστε και εσεί και εμεί να προχωρήσουμε στι επιτροπέ μα. Δεδομένου ε, πρέπει κάποια πράγματα που ε, από νομοθετική πλευρά έχουν ήδη αποφασιστεί να τα κλείσουμε Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συνεισηγητές. Τρία λεπτά στον καθένα. Ποιος θέλει να αρχίσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της Επιτροπής ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ που κατέθεσαν τροπολογίες, όπως ε, είπατε, σχεδόν έχουμε χίλιες τροπολογίες και έχουμε και τις ε, γνωμοδοτήσεις άλλων τεσσάρων επιτροπιών. Μαζί με τους άλλους συνεισηγητές και τους ε, συγητές έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε για την σύνταξη των συμβιβαστικών τροπολογιών. Ξέρουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Είπαμε ότι θα ψηφίσουμε εμείς 4 Μαρτίου και δεδομένου ότι πρόκειται για ένα μηχανισμό πολύ πολύπλοκο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε ε, σε κάποια συμπεράσματα τα οποία ελπίζουμε ότι θα τύχουν της έγκρισης από πολύ μεγάλο αριθμό συναδέλφων. Βεβαίως είμαστε ανοιχτοί σε ε, κάποιες ε, προτάσεις που θα κάνουν συνάδελφοι, αλλά ε, μας, μας είναι ιδιαίτερα προσφυλή συλλογική της όλης έκθεσης. Βλέπουμε ότι έχουν κάποιες τροπολογίες ε, από δημιουργήσει μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν οδηγήσει μεγάλες συζητήσεις εκ μέρους μας. Τώρα, το να μπορέσουν ε, αυτοί οι δύο μηχανισμοί να ε, αποτελέσουν έναν ε, κοινό μηχανισμό είναι κάτι το οποίο υπάρχει σε κάποιες τροπολογίες, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο εμεί ιδιαιτέρως Θέλουμε όμως όλα αυτά τα θέματα να αντικατοπτρίζονται σωστά στα στους δημοσιονομικούς μηχανισμούς. Τώρα, όσον αφορά τη διακυβέρνηση, είναι πάρα πολύ διαρθωμένος ο τρόπος με τον οποίο πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε ε, να δημιουργήσουμε συστήματα προστασίας ώστε να μπορέσει για την καθαρισμό των πολιτικών να έχει ε, σημασία αυτό το οποίο θα πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων με εμπεριστατωμένη συζήτηση για, για τις... Ε, Επίση, πράξεις. Επίσης, υπάρχουν ε, κάποιες τροπολογίες που αλλάζουν ε, την ε, λογική όσον αφορά κάποια θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας. Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να είμαστε ρεαλιστές και να μην ε, γίνει πολύ ο μηχανισμός, διότι θα χαθεί η ιδέα της ευελιξίας και δύο λόγια για τον προπολογισμό που είναι σημαντικός. Οι δικές μας προτάσεις πρέπει να πω ότι λαμβάνουν υπόψη την παρούσα κατάσταση των κονδυλίων που προβλέπονται για τις διάφορες ε, γεωγραφικές ζώνες και για τα διάφορα θέματα και έχουμε κάνει προβολές για την επόμενη μουσιονομική περίοδο λαμβάνοντας υπόψη για το MFF ε, για, το, ε, για PDP δηλαδή, ποιες είναι οι προτινόμενες, τα προτινόμενα ποσά. Θέλουμε να διατηρήσουμε τα ποσά που υπάρχουν και την ευελιξία στα πλαίσια αυτού του νέου μηχανισμού. Βεβαίως είμαι ανοιχτός σε διάλογο και σε εξέβρεση λύση με τους άλλους συναδέλφους ώστε να παρουσιάσουμε μια πολύ ισοσκελισμένη πρόταση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, Κριστιά. Μετά από τον Κριστιάν, ποιο θέλει να λάβει το λόγο, ο κύριο Παντζέρη. Grazie, molto brevemente, anche perché... Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Βεβαίω και συμφωνώ με τα όσα είπε ο Κριστιαν Ευχαριστώ πολύ τους ε, συναδέλφους που κατάθεσαν τροπολογίες. Αυτό αποδεικνύει και το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει συγκεντρώσει αυτός ο κανονισμός, ο νέος κανονισμός. Θα ε, μιλήσω περισσότερο για τα θέματα που αφορούν τις ε, τροπολογίες στο μεγαλύτερο ποσοστό. Τους ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν είναι οι τομείς ισότητα των φύλων, δικαιώματα των νέων, των παιδιών, είναι προτεραιότητες των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδιώκουμε λοιπόν την ενίσχυση των τομέων αυτών μέσα από τις τροπολογίες που θα προσδιορίσουμε. Επίσης η νέα διαδικασία που σας προτείνουν τα συνεισηγητές σας για την ε, άρση τη ε, στήριξη υπέρ των των δικαιωμάτων έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Στο άρθρο 23, παραδείγματι, έχουμε μια, έχουμε μια σειρά από τροπολογίε που στόχο έχουν την ενίσχυση και προστασία του ρόλου των ε, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, που πιστεύω θα είναι και ο καλύτερο τρόπο να προσφέρουμε ουσιαστική βοήθεια σε όποιους κινδυνεύουν. Στο άρθρο 32 επίσης αξιολόγηση. Θα δείτε μια σειρά από τροπολογίες που ζητούν τη συμπερίληψη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού. Και νομίζω ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι εγχώριες, είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθούν. Ειδικά για τον τομέα των ανθρωπινών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Αυτά. Ευχαριστώ όλους ε, τους συναδελφούς που συνεργάστηκαν στη δουλειά αυτή. Η δουλειά μας κράτησε αρκετού μήνες. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί βεβαίω, Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να στεφθεί με μια επιτυχή ολοκλήρωση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. κέρενς Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το έργο που αναλάβαμε ως συνεισηγητές μόνο ε, έργο ρουτίνας δεν είναι. Είναι τόσο σημαντικές οι προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εξωτερικές της σχέσεις, για τις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι οι εταίροι και παραλήπτες, αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί έχουμε και τα δικά μας προνόμια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δικές μας αρμοδιότητες. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη όταν αναλύουμε λοιπόν αυτό το σχέδιο έκθεσης. Και το σχέδιο αυτό έκθεσης όπως το έχουμε διαμορφώσει ως συνεισηγητές, αν εγκριθεί θα ε, πληρώσει ένα σημαντικό ε, δημοκρατικό έλλειμμα. Με τη συμπερίληψη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη στον προπολογισμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει, αν μη τι άλλο, ένα σημαντικό προνόμιο. Κάτι που είναι εύλογο και το έχουν όλα τα εθνικά κοινοβούλια που αποφασίζουν για τις δαπάνες. Νομίζω ότι έτσι θα τεθεί ε, τέρμασε κάτι αναχρονιστικό και παροχημένο, ένα δημοκρατικό έλλειμμα που μας βασανίζει από την αρχή της ύπαρξής μας. Δεύτερον, για τη διακυβέρνηση. Δεν θα πρέπει να κάνουμε κατάχρηση της δυνατότητάς μας ε, να ε, χρησιμοποιούμε παντού τις κατεξοδότηση πράξεις και παράλληλα ως συνεισηγητές προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφύγουμε αυτόν τον πληθωρισμό κατά εξοδότηση πράξεων. Δεν θέλουμε, είπαμε, να σας εμποδίσουμε να πελαγοδρομήσετε, αλλά ούτε και εσείς πρέπει να μας εμποδίσετε στον προγραμματισμό μας και στον καθορισμό στρατηγικών προτεραιοτήτων. Θέλουμε να έχουμε λόγο. Και αυτή είναι η εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις πρώτες εκλογές του 1979. Και το έχουμε επισημάνει για όσο περισσότερε αρμοδιότητε έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο περισσότερε ευθύνε αναλαμβάνει, τόσο πιο υπεύθυνο πρέπει να γίνεται. Και γι' αυτό δεν έχουμε τις εκτελεστικές ε, πράξεις. Αυτό που θέλουμε να, είναι να έχουμε λόγο για τις ε, στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά θέλουμε να είμαστε το αντίβαρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είμαστε όχι μόνο αντίβαρο, αλλά και σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί έχουμε πολλά κοινά. Και γι' αυτό, για τον προϋπολογισμό, για τις πιστώσεις και τα κονδύλια, ε, καλό να γίνουν κάποιες αλλαγές υπό το πρίσμα των κοινοβουλευτικών προτεραιοτήτων. Γιατί λοιπόν μειώσαμε το αποθεματικό, το μειώσαμε, γιατί κρίνουμε ότι 10,2 δισεκατομμύρια στο αποθεματικό είναι υπέρογκο ποσό. Αυτή είναι η γνώμη μας. Και το μειώσαμε κατά 50%, όχι κατά 50% όπως ήθελα εγώ. Τελικά συμφωνήσαμε οι συνεισηγητέ στα 7,5 δισεκατομμύρια. Πιστεύουμε ότι αρκεί αυτό το ποσό για το αποθεματικό. Επίσης έχουμε μια δεύτερη ασφαλιστική δικλίδα, ε, ώστε η ευελιξία να μην δίνει λευκό επιταγή στην εκτελεστική εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και προσθέσαμε τις κατεξοδότηση πράξεις. Επίσης φροντίσαμε ώστε να μην τα βλέπουμε όλα από τη σκοπιά της μαθηματικής ακρίβειας. Δεν μπορούμε πάντα με την εξονυχιστική λεπτομέρεια να προβλέπουμε ποιε θα είναι οι δαπάνες μας για το φύλλο, για την ισότητα των φύλων. Αυτό είναι περί τη συζήτηση. θέλουμε μια αγνήσια πολιτική εξισορρόπησης και ισότητας των φύλων, θέλουμε μια οριζόντια προσέγγιση συνεκτίμησης του διάσταση φίλου που θα χαρακτηρίζει όλες τις συζητήσεις και όλα τα σχέδια της Επιτροπής. Είτε χτίζουμε σχολείο, είτε νοσοκομείο, οποιαδήποτε άλλη υποδομή, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φίλου και της δικαιοσύνης ε, και της εις μεταχείρισης των φύλων. Να πω δύο λόγια και για το κλίμα. Έχουμε αφενός τη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν το 25%, των αναπτυξιακών προγραμμάτων που θα πρέπει να αφιερώνονται στο κλίμα, κατά μέσο όρο, εμείς το αυξήσαμε αυτό το ποσοστό στο 30%. Μάλιστα κάποιος τροπολογής ζήτησε μέχρι 50% των αναπτυξιακών κονδυλίων να πάει στο κλίμα. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ζήτησε 30%. Εμείς εκεί ε, περιοριστήκαμε στο 30%. Και θα σας πω γιατί δεν προτείναμε υψηλότερο ποσοστό, γιατί λέγαμε ανέκαθεν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι προβλήματα που ε, προκλήθηκαν από αυτούς που μόλυναν το κλίμα, από εμά δηλαδή. Εμείς ε, ρυπάναμε το κλίμα, οπότε έχουμε ένα χρέος προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Οπότε αυτά τα κονδύλια για να εξηλωθούμε από την υποχρέωσή μας θα πρέπει να είναι επιπλέον κονδύλια. Και βλέπω ότι αυτή η επιχειρηματολογία στην πορεία εξαφανίστηκε, ενώ ήταν ανέκαθεν μια διεκδίκηση δική μας. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι και για τη μέθοδο εργασίας μας. Και θα ήθελα να πω εκ μέρους και των τεσσάρων συνεισηγητών ότι έχουμε δύο ομάδες από ε, τις δύο επιτροπές, ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ, πολύ αξιόλογους συνεργάτες, πολύ αφοσιωμένους εξαιρετικούς επαγγελματίες και έχουμε πραγματικά μεγάλη ευγνωμοσύνη νιώθουμε προς τα δύο αυτά επιτελεία και πραγματικά θα μας καλομάθουν σε τέτοιο άρτιο έργο και συνεργασία. Ευχαριστώ αυτά. Ευχαριστώ κύριε Γκέρενς. Ο Φρανκ Έγγελ δεν είναι εδώ. Σας άφησε λοιπόν και το δικό του χρόνο ομιλίας. Και έτσι εξισορροπήσαμε την εκπροσώπηση της ΑΦΕΤ και της ΔΕΒΕ. Ανταλλαγή απόψεων. Έχουν ζητήσει αρκετοί σκιώδεις και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο. Ο κύριος Νόιζερ πρώτος. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ και πολύ σύντομα για να εκθέσω τη θέση, τις θέσεις μας ως ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών για την Επιτροπή της Ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, 0,7 ο στόχος που καταγράφεται, 0,2% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Το έχουμε στην πρόταση ήδη. Νομίζω ωστόσο ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες Ξέρω ότι είναι σαφής η κατάσταση για ορισμένε χώρες, η Ινδία όμως, η Βραζιλία. Πρέπει να έχουν διαφορετική μεταχείριση από τις λιγότερο ανεπτυγμένε χώρες. Στην κλιματική αλλαγή, στο θέμα της ισότιμη μεταχείριση των φύλων, έχουμε προχωρήσει σημαντικά στις προτάσει των εισηγητών. 50% στην κλιματική αλλαγή ζητούμε. Και αυτό δεν σημαίνει μόνο έργα ή σχέδια για την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής, αλλά και έργα και σχέδια της βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, στην ε, δε ισότητα των φύλων έχουμε 20%. Ε, η έννοια αξιοπρεπής θέση εργασία θέλουμε να συμπεριληφθεί στην έκθεση, όχι μόνο προδιαγραφέ Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω λέγεται ήδη στην έκθεση, αλλά στο πεδίο τη ανάπτυξη θέλουμε να είναι η αξιοπρεπής θέση εργασία, μια σαφή έννοια, που θέλουμε να εξασφαλίζονται και να υλοποιούνται με μια ευρωπαϊκή εγγύηση. Τελευταία παρατήρηση. η ποσοτική αξιολόγηση της ασφάλειας, η στάθμιση της ασφάλειας σε σχέση με την ανάπτυξη, γιατί δεν έχουμε προβλημό προς την επιδίωξη της, ασφάλειας, της μέσω των αστυνομικών δυνάμεων, αλλά όταν μιλούμε για στρατιωτικές δυνάμεις είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι αυτές χρειάζονται για την υποστήριξη της ανάπτυξης. Χρειάζονται άλλα μέσα, λοιπόν. Ναι, ασφάλεια χρειάζεται, αλλά με άλλα μέσα. Ευχαριστώ, Νόρμπερτ. Τσάλ Στάνακ, δύο λεπτά. Δεν σκοπεύω να λάβω το λόγο μια και μίλησα την προηγούμενη φορά, αλλά η ομάδα μου υποστηρίζει πλήρως την πρόταση με τα νέα μέσα για την αναπτυξιακή συνεργασία. Πιστεύουμε ότι θα προσφέρουν περισσότερη ευελιξία, οικονομία κλίμακος. Επιφυλάξει έχουμε για τη γειτονία, για το αν θα πρέπει να περιλαμβάνεται και αυτή αλλά δεν έχει κατασταλάξει ακόμη στη τελική της θέση η ομάδα μου. Εν πάση περιπτώσει όμως γενικά την ιδέα ότι επιδιώκεται η οικονομία κλίμακος με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουμε στις ε, διάφορες περιοχές και την ευέλικτη αξιοποίηση των ε, πόρων από τον προϋπολογισμό την ε, καλωσορίζουμε βέβαια η νέα επιτροπή μετά τις εκλογές δεν είναι εκείνη που θα πρέπει να την υλοποιήσει αλλά πρέπει το νομοθετικό πλαίσιο να έχει ολοκληρωθεί πριν από την ε, αφιπηρέτηση του Κοινοβουλίου κάποιες τροπολογίες θα καταθέσουμε και εμείς σε αυτό το χρόνο ο Πρόεδρος ευχαριστώ κυρία Σαρχεντίνη ευχαριστώ Πρόεδρε Είχαμε στην Επιστροπή Ανάπτυξη επίσκεψη του ΟΣΑ με μια ε, αξιολόγηση από ισοτήμους ε, του Ντάκ του εγγράφου προς ε, επιβεβαίωση των δαπανών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 55 μόνο των οποίων πάνε στις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Εάν κοιτάξετε λοιπόν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με το αναπτυξιακό ταμείο η κατάσταση μπορεί να είναι διαφορετική και, είναι διατεθειμένοι από ό,τι φαίνεται να το περιλάβουν και αυτό, αλλά δεν ξέρουμε εάν θα πραγματοποιηθεί στο τέλος και αυτή η συμπερίληψη εν ώψη του ΝΤΑΣ Τι θα γίνει λοιπόν σε μια μεταγενέστερη φάση, αν αργότερα πει το Συμβούλιο ότι δεν είναι διατεθειμένο να υπολογίσει μέσα στις δαπάνες αυτές το αναπτυξιακό ταμείο. Το μαξιλάρι νομίζουμε ότι είναι υπερβολικό, δεν είναι απαραίτητα ε, υποφελής για τις αναπτυσσόμενες χώρες η ευελιξία, το μαξιλάρι δεν είναι κάτι το προβλέψιμο. Εμείς θέλουμε κάτι το προβλέψιμο. Έτσι λοιπόν θεματικοί πυλώνες που θα εξασφαλίζουν πως οι δαπάνες όντως πηγαίνουν στις προτεραιότητες έχουν ε, τεράστια σημασία. 50% για την κλιματική αλλαγή. Αυτό οπωσδήποτε πρέπει να είναι στόχος μας. Επίσης, μικρότερα ταμεία. Η χρηματοδότηση κατά εξουσιοδότηση μπορεί να είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει στην αξιοποίηση κονδυλίων κατά τρόπο ταχύ και στοχευμένο στην κοινωνία των πολιτών για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα. Επίσης, άρθρο 3, στόχοι στόχοι που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τα άρθρα τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα το 208, που αναφέρεται πω στο σύνολό τη η εξωτερική μα πολιτική πρέπει να στοχεύει σε μια βιώσιμη ε, απάλληψη τη ε, φτώχεια. Κάτι ακόμα, Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή οργανώνουμε τη δική μας διαπραγματευτική εντολή και άρα δεν χρειάζεται να παρακολουθούμε τα ευχολόγια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μπαίνουμε στη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό θα ακολουθήσει αργότερα. Αυτή τη στιγμή αυτό που είναι απαραίτητο είναι να έχουμε μια πολύ σαφή και φιλόδοξη διαπραγματευτική εντολή. Εν τίτσι είπατε έτσι το λέμε, έτσι το βαφτίσαμε το μωρό. Το άκουσα αλλά δεν το πίστεψα. Εντάξει, εγώ νόμιζα ότι ήταν NDICI, αλλά εσείς το προφέρετε NDC. Πολύ καλά. NDC. Η κυρία Λέζινγκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολλές οι τροπολογίες εκ μέρους Ευρω... της ε, ΓΚΟΕ. Μπορώ να πω ότι 80% των τροπολογιών αυτών μπορούμε να τις ε, υποστηρίξουμε. Ωστόσο, αποφασιστικά καθόμαστε κατά της αναφοράς και ε, συμπερίληψης της δραστηριότητας στρατιωτικών παραγόντων και ιδιαίτερα όσον αφορά την αξιοποίηση ανατοξιακών κονδυλίων που θα μπορούσαν να πάνε σε λεγόμενους στρατούς εταίρους. Και το CPST επίσης, μέτρα του CPST. Γιατί αν υπενθυμίσουμε ότι Ε, θεσπίζεται και το μέσον για την ειρήνη στην Αφρικά, υπάρχει ο κίνδυνος της ε, ε, παρέκκλησης και της διολίστησης από τους πολιτικούς στόχους τους στρατιωτικούς και να εξυπηρετηθούν αυτοί από την αναπτυξιακή μας πολιτική. Επίσης, ο μηχανισμός ταχείας ανταπόκρισης όπως αναφέρεται στο κείμενο στο σημείο C η διεύρυνσή του λοιπόν σε ε, αντιμετώπιση εξελίξεων και προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής σημαίνει ότι αδίποτε, οδηποτε τομέας εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να θεωρηθεί τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμε το μηχανισμό ταχείας αντίδρασης. Εάν ε, μείνουμε λοιπόν στην πρόταση Επιτροπής, τότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλη προσπάθεια, γιατί αυτή, να συστήσουμε τίποτα περισσότερο, γιατί αυτός ο ορισμός μπορεί να περιλάβει τα πάντα. Και εν τέλει, για τα μέσα δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε προτείνει. Ερωτώ μόνο ποια είναι η λογική που οδήγησε τους εισηγητές να μην περιλάβουν στο κείμενο της έκθεσης την διεκδίκηση για χωριστά μέσα και να την προβλέψουν μόνο για τον τριμερή διάλογο. Περιμένω απάντηση. Ο Μίχελ Γκάλερ είναι Ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι ξεκινώντας καλή δύναμη σε αυτήν την ε, διελκυστίνδα στους συνσηγητές μας. Ελπίζω ότι θα ευοδοθεί η προσπάθεια. και στη τελική φάση με το Συμβούλιο. Δεν έχω ακούσει απάντηση από τους ηγητές ε, στο ερώτημά μου. Εγώ έχω διατυπώσει πέντε τροπολογίες για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είναι σε equal footing, όπως λέμε, δηλαδή ισότιμη βάση η προαγωγή της δημοκρατίας με του αγώνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώ μπορούμε λοιπόν αυτά να τα εξασφαλίσουμε σε ισότιμο επίπεδο, να μην προάγουμε μόνο ανθρώπινα δικαιώματα, να μην υποστηρίζουμε μόνο την κοινωνία των πολιτών που ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και να ε, βοηθήσουμε στα επόμενα βήματα στην προαγωγή τη δημοκρατία. Νομίζω ότι το ευρωπαϊκό καταπίστευμα για τη δημοκρατία πρέπει να έχει καλύτερε πιθανότητε επιτυχία. Επίσης, η Ρεβέκα Χάρμς ε, έθεσε ένα άλλο ερώτημα που με απασχολεί και εμένα. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε θεσμικό επίπεδο να υποστηρίζει την ε, παρατήρηση εκλογών, που μερικές φορές ακόμα γίνεται ad hoc με συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένα έργα δηλαδή, αλλά πιστεύω ότι πρέπει και δεδομένου ότι έπονται εκλογές να είμαστε έτοιμοι να αναπτύσσουμε τις δραστηριότητες ε, επιτήρησης, ε, παρατήρησης των εκλογών. Δεν άκουσα για τις λεπτομέρειες αυτές τις θέσεις, των, η παρατήρηση από πλευράς των ε, Θα ήθελα να ακούσω κάποιες έστω ενδείξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ. Ε, ο κύριος Χάνη είναι επόμενος ομιλητής. Πολύ σύντομα. Εκπροσωπώ την κυρία Κλέρ Μούντι που κολλείται σήμερα. Είναι μεγάλο τιμά τη νομοθεσία μα να αφήσουμε το στίγμα μας στο παγκόσμιο προσκήνιο, έξω και ο τεράστιο αριθμό τροπολογιών. Κάνουμε πολλά στον τομέα αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμη περισσότερο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε κάποιε δράσει ε, ε, στη Σρι Λάνκα, γιατί δεν ε, είναι επιλέξιμο το πρόγραμμα. Οπότε η αποτροποποίηση ε, του Μηχανισμού Γειτονίας Ανάπτυξης θα πρέπει να λάβει υπόψη τις αλλαγές στο, στους δύο πυλώνες και όπως είδαμε και στον Τομπά, σίγουρα η αποναρκοθέτηση θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τα αναπτυξιακά κονδύλια. Επίσης, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βγει από τους γεωγραφικούς ή θεματικούς πυλώνες για να καταφέρουμε να απαλλάξουμε τον κόσμο, τον πλανήτη από τις συνάρκες στο μέλλον. Ευχαριστώ. Εξαντλήσαμε τον κατάλογο των ομιλητών, οπότε θα δώσω τώρα το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Βεσά Γκριμπό, που είστε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Γκριμπό από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, Αναπτυξιακή Συνεργασία Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το έργο των συνεισηγητών του και για την ταχύτητα και την ποιότητα, την ερτιότητα αυτού του έργου που επέτρεψε ε, την ποιοτική σήμερα συζήτηση ενώπιση της υιοθέτησης από κρυστάλλου στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είδαμε την πορεία Έχω πάρει συζητήσει μετά και τι τροπολογίε πάντω κατά την γνώμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε μια τεράστια ευκαιρία να βελτιώσουμε τη χρηματοδότηση των εξωτερικών δράσεων τη Ένωση και σημαντική ευκαιρία να ενισχύσουμε τη δημοκρατία στι εξωτερικέ μα δράσει και κυρίω μέσω τη ενσωμάτωση στον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη. Ακούσαμε σήμερα τον εκπρόσωπο τη Ρουμανική Προεδρία. Πιστεύω ότι ε, θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκεί πλήρω το ρόλο του. Γιατί είναι μια απόφαση που θα πρέπει να λάβουμε το Συμβούλιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από αυτήν την άποψη η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη. Επίση, ε, ε, οι ανησυχίε που εκφράσατε για τη διακυβέρνηση είναι ευλόγε και θα ληφθούν υπόψη. Ε, με ξεχνάτε ότι μεγάλος αριθμός κατεξοδότηση πράξεων είναι υπερβολικός, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ελαστική εφαρμογή του ε, μηχανισμού, γιατί θα προσκρούσουμε με τις πολλές κατευθυντές πράξεις θεσμικές και άλλες δυσκολίες και δεδομένου του χρόνου που χρειάζεται, δεδομένης αρχής εταιρική σχέσης, της τροφοδότησης των εταίρων μας, αλλά και των κοινών αποστολών. Παρ' όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να συνεχίσει τη συζήτηση για να βελτιώσει την κατάσταση και να εξασφαλίσει ε, με διακυβέρνηση του μηχανισμού που θα ανταποκρίνεται στι προσδοκίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα συνεχιστεί τι επόμενε εβδομάδε συζήτηση για να εντοπίσουμε τα κοινά μα σημεία και που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Τρίτον, θα ήθελα να επανέλθω ε, στους διάφορους στόχους μας. Καταρχήν, το θέμα της επιλεξιμότητα ε, δημόσια βοήθεια και δαπάνε. 92% είναι το κατόφλι που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολύ πιο φιλόδοξο από το ισχύον. το 95% ή άλλο ψηλότερο ποσοστό θα δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση κάποιων δαπανών, γιατί ο συγκεκριμένο μηχανισμό αντικαθιστά περίπου 10 άλλου μηχανισμού και καλύπτει και την συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες και πολλά άλλα σημεία συνεργασίας που ίσως δεν είναι επιλέξιμα από τον μηχανισμό σε θέματα ασφάλειας για παράδειγμα, αλλά ο μηχανισμός είναι κυρίως αναπτυξιακό μέσο και αυτό φαίνεται με το κατόφλι. Αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται ένα περιθώριο λιγμών για να μην δημιουργήσουμε περιτά προβλήματα στην εφαρμογή αυτού του μηχανισμού. Γειτονία ανάπτυξη και διεθνού συνεργασία. Επίσης, όπως είπαμε πολύ προαναλύσαντες, δεν θα πρέπει να υπερφορτώνουμε τους στόχους μας για να μην γίνει ένας κλειός άκαμπτος αυτός ο μηχανισμός και άκαμπτη παροχή ενίσχυσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν, μια και έχουμε αρκετούς στόχους, να μην προσθέσουμε και νέους. Θέλουμε φιλόδοξους και ρεαλιστικούς στόχους για να μην είναι αντιπαραγωγικό τελικά το αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους κονδύλια, ε, είναι απαραίτητο αρκετό αποθεματικό. Τα 10 δισεκατομμύρια είναι πολύ λιγότερο από το τμήμα του ΦΕΔ, του Ταμείου Ανάπτυξης για το αποθεματικό, οπότε ε, στα 90 δις να έχουμε 10 δις αποθεματικό δεν είναι υπερβολικό κατά τη γνώμη μας, είναι το ελάχιστο απαραίτητο. Βέβαια είναι αυτονότητα ότι θα συζητήσουμε τον τρόπο διαχείρισης του θεματικού, αποθεματικού και το ρόλο των διαφορών εταίρων. Επίσης είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε αυτό το ποσό και για το τρίτο πυλώνα τη άμεση αντίδραση που εξ ορισμού θα πρέπει να είναι φωτιασμένος με αρκετά κονδύλια για να αντιμετωπίσουμε προσδόκητες ε, ε, κρίσει. Και από το προηγούμενο πι ε, διδαχθήκαμε να έχουμε μεγάλο περιθώριο λιγμών για να αντιμετωπίσουμε τις απρόσμενες εξελίξεις. Επίσης, επιμένω στην ανάγκη της, της ε, αναγνώρισης της σημασίας των επενδύσεων, του κεφαλαίου των επενδύσεων. Και μάλιστα φάνηκε αυτό και από την συζήτηση με τον ΩΣΑ. Και έχουμε ενισχυμένη τα συμμετοχή της Επιτροπής ΕΤΕΠ, της, Επιτροπής, της Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ. Από την Digineer, η κυρία Αναπήρες, η επόμενη ομιλητρία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κι εγώ, όπως και ο Βενσάν, να σας ευχαριστήσω για την έκθεση και κυρίως το πόσο πολύ προσέχει το θέμα αυτό που φοράει τη Γετανία. Υπάρχουν στοιχεία της ε, έκθεση της Επιτροπής στην έκθεση αυτή και κάποιοι από τους ε, συνεισηγητές αναφέρθηκαν στα θέματα αυτά. Απ' τη μια, ο μηχανισμός αυτός προσφέρει ασφαλή και καλύτερη χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τις της σχέσεις μας με τις χώρες γειτονίας και απ' την άλλη διασφαλίζει το στοιχείο της διαφοροποίησης που μας επιτρέπει να έχουμε μία γειτονία, όχι μία γειτονία όπως λέγεται Ανατολάς και μία στο Νότο. Θέλουμε αυτή την ευελιξία την οποία έχουμε στο μηχανισμό αυτό να συνεχίσουμε να την έχουμε, τον έχουμε και τον έχουμε και μία νέα γειτονία. Στο δεύτερο μέρος θα θέλαμε να επιμείνουμε στο εξή τώρα. Όντως, υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι όπως ελέγχθηκε. Άκουσα κάποια σχόλια που είπαν κάποιοι συναδελφοί σα ότι θα πρέπει να ε, μπορεί να προγραμματιστεί. Το γεγονός όμως είναι ότι Έχουμε έρευνε που λέγουν ότι θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία και περισσότερου σπόρου σε περίπτωση συμπληρωματική κρίση. Θα πρέπει λοιπόν αυτή την συμπληρωματική ευελιξία στην πρόταση να την διατηρήσουμε κυρίω για την γειτονία για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που ενδεχομένω θα παρουσιαστούν. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτά τα στοιχεία να τα διατηρήσουμε. Και δύο πολύ σύντομε παρατηρήσει για κάποιε ειδικέ τροπολογίε. όσον αφορά του ειδικού στόχου τη γειτονία, που είναι κάτι το οποίο και εμεί συμμεριζόμαστε. Πρέπει να δούμε την αναθεωρημένη πολιτική γειτονία και να δούμε αν μπορούμε να αντικατοπίσουμε το γεγονός ότι η κύρια πολιτική προτεραιότητα είναι σταθερότητα. Αυτό στο στοιχείο. Και δεύτερον, όσον αφορά την ε, προσέγγιση βάση επιδόσεων, όπως είπε και ο Βενσό θα πρέπει να σας πω ότι αυτή, αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερο εδώ είναι ότι θα πρέπει να εκτιμηθούν πάρα πολλά ποιοτικά κριτήρια. Άρα δεν πιστεύουμε ότι ο τρόπος αυτός που ε, αναφέρανε, ανέφεραν κάποιοι συναδελφοί σα με πράξεις εξουσιοδότηση είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Ε, ευχαριστώ κυρία Πύρες. Τελικά ο κύριος Γιώργη Μίλλερ από την... Ε, α, η Μαρή Λόρντεμπαρ από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ Σα ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση αυτή και για το ενδιαφέρον που επιδείξατε για τον μηχανισμό αυτό της γειτονίας και για την ε, διεθνή συνεργασία. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω τέσσερα σημεία. Πρώτα απ' όλα, σημειώνουμε με θετικό τρόπο ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη όσον αφορά την πρόταση, όσον αφορά τη δομή δηλαδή. Να έχουμε ένα σφαιρικό μηχανισμό στον οποίο θα υπάρχουν και η ιδιαιτερότητα της πολιτικής μας όσον αφορά τα θέματα γειτονίας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Υποστηρίζουμε βεβαίως και αυτό που λέγεται ότι θα πρέπει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου να συμπεριληφθούν τα κονδύλια στον προϋπολογισμό και να υπολογιστούν. Δεύτερον, θέλω να υπενθυμίσω ότι ο στόχος της πρότασης αυτή είναι να μπορέσουμε να θεσπίσουμε ένα μηχανισμό που θα μπορεί να υποστηρίζει περισσότερο την πολιτική που θέλουμε να κάνουμε σε πλαίσιο ανάπτυξης εξωτερικής βοήθειας και η ευελιξία είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορούμε να αντιδρούμε έγκαιρα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ένα αποθεματικό σε θέματα συνεργασίας και ανάπτυξη είναι απαραίτητα. Άρα είναι σημαντικό να διατηρήσουμε ένα σημαντικό περιθώριο ε, ελιγμών όσον αφορά κάποια κονδύλια τα οποία μπορούμε να διαθέσουμε όπως θέλουμε και να διατηρήσουμε και κάποια κονδύλια σε περίπτωση ταχείας αντίδρασης εκ μέρους μας. Δείτε, αυτό είναι σημαντικό για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τρίτη παρατήρηση όσον αφορά τους στόχους. Σημειώνοντας με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις που έγιναν όσον αφορά τους επιμέρους αντικειμενικούς στόχους. Θέλω να υπενθυμίσω το ότι εάν ε, προβλέψουμε πάρα πολλούς επιμέρους στόχους, θα μειώσουμε την ευελιξία. Και κυρίως Γκέρενς. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αυνοήσουμε το διάλογο με τις ε, χώρες τι οποίες έχουμε τέτοιου εταιρική σχέση. Τελευταία παρατήρηση όσον αφορά την διακυβέρνηση. βεβαίως με μεγάλο ενδιαφέρον λαμβάνουμε υπόψη τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι θα πρέπει παρόλα αυτά να ακολουθήσουμε μία διαδικασία προγραμματισμού, ώστε να είμαστε σε θέση να δίδουμε πιο έγκαιρα και με πιο ευέλικτο τρόπο ε, απαντήσεις και να ανταποκρινόμαστε στις ε, καταστάσεις ίσως και τελευταίας στιγμής. Ευχαριστώ. Από την Επιτροπή κάποιος άλλος, από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, όχι. Ποιος ακολουθεί παρακαλώ, ποιος θα λάβει το λόγο από τους συγκητές. κύριε Γκέρενς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και θα ήθελα να λάβω το λόγο σε κάποια σημεία σημαντικά πιστεύω καταρχάς για το εγκληματική αλλαγή ας μην ε, διαφωνήσουμε για τα ποσά ε, πριν αναλυφθεί δηλαδή μια οριστική απόφαση θα ήθελα η Επιτροπή να μας ενημερώσει για τον απολογισμό των 100 δισεκατομμυρίων που είχαν, δοθεί, που είχαν χορηγηθεί ως υπόσχεση στο Παρίσι. Αυτά τα 100 δισεκατομμύρια λοιπόν από πού θα προκύψουν, πώς θα χρηματοδοτηθούν και δεύτερον πώς θα καταρμηθούν. Να μην έχουμε διπλό κενό. Ό,τι είναι να καλυφθεί σαν έξοδο από τα 100 αυτά δισεκατομμύρια να μην χρειάζεται να καλυφθεί από το NDICI. Για τον κύριο Νόιζερ και τις αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι έχουμε την επιλογή μεταξύ δύο ε, διαφορετικών διατυπώσεων η μία που ορίζει πως θα πρέπει ε, στην εξωτερική μας δράση να τηρούμε την προ... τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Οπότε θεωρούμε ότι με βάση αυτά τα πρότυπα είναι και η θέση εργασίας αξιοπρεπής και άρα ακολουθούμε τις ε, συστάσεις του ILO. Και τρίτον, εκεί που αναφέρεται σε μια ανάμειξη της πολιτικής ασφάλειας και της ανάπτυξης ο Νόρμπερτ Νόιζερ. Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που δεν μπαίνουν στο NDICI με παρέμβαση στρατιωτική όπως μέσω, μέσω της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που είναι εκτός του NDICI και της ευρωπαϊκής διευκόλυνσης για την ειρήνη που είναι πάλι εκτός προπολογισμού. Ας δούμε λοιπόν ε, τι πόσα θα δαπανηθούν μέσα από αυτούς τους διάβλους και να δούμε μετά εάν ε, έχουμε φορτώσει πολύ το εργαλείο μας με θέματα συναφή με τη στρατιωτική ασφάλεια, με το στρατιωτικό σκέλος, σκέλος της ασφάλειας. Ο Τσάλς Τάνακ, που δεν είναι εδώ. Προτιμά μας είπε ε, τον αποχωρισμό της πολιτικής γειτονίας από το μέσον αυτό. Δεν είναι μόνος, δεν είναι ο μόνος ε, και εμείς ε, οι συνεισηγητές αυτό θέλαμε, αλλά καταλήξαμε τελικά στην πρόταση που βλέπετε. Διακυβέρνηση. Κατά υψηδότηση πράξης. Επαναλαμβάνω πως δεν υπερβάλαμε, δεν διατυπώσαμε ακραίες προτάσεις στο πλαίσιο όμως της Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης εκδηλώνεται μια αλλεργία νέα, ακόμα μεγαλύτερη του κ. Φλερ με το που βλέπει κατά το τη συμπράξη, βλέπουμε τα αντισώματά του να παίρνουν μπρο. Για να μην πω αλλεργία, σχεδόν γενικευμένη απόρριψη από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για νεωστή φορά, λοιπόν, παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την ε, θέση και τις προνομίες και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα στην προοπτική αυτή. Ε, δεν ήμασταν εξ αρχής στο επίπεδο αυτό. Καταλήξαμε σε συμβαστικές λύσεις που επιτρέπουν πάντως ε, βήμα το βήμα να ε, παγιωθούν και να επιβεβαιωθούν οι προνομίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό θεωρώ ότι και το Συμβούλιο θα μπορέσει να συμφωνήσει στην έγγραφη στον προπολογισμό του Ταμείου για την Ανάπτυξη. Δεν θα πάμε να δώσουμε μαθήματα δημοκρατία σε όλε τι χώρε τη Αφρική ενώ και να του λέμε ότι τα κοινοβούλια του πρέπει να, περι... συμμετέχουν περισσότερο στο δημοκρατικό γίγνεσθε όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει λόγο για το σχετικό ταμείο. Νομίζω ότι είναι η ευκαιρία να βάλουμε ένα τέλο σε αυτήν την ιστορία. Που είναι και ένα χρονισμό. Ευχαριστώ και ελπίζω να κάλυψα όλε τι ερωτήσει που με αφορούσαν. Ο πρόεδρο ερώτησε. Ο Κριστιαν ο Πιερ Αντώνιο. Ξέρω ότι δεν έχουμε παραπάνω από τις 6 και 30 ακριβώς. Επομένως από δύο λεπτά ο καθένας, Κριστιαν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίχαλ Γκάλερ έκανε κάποιες ερωτήσεις οι τέσσερις συνεισηγητές έχουν συμφωνήσει επί της αρχής, δεν έχουν λάβει απόφαση, αλλά έχουμε αποφασίσει από 10 δισεκατομμύρια να πάμε στα 7,5 δις στο αποθεματικό, αλλά απ' την άλλη δεν θέλουμε να κάνουμε άκαμπτη τη ρύθμιση με την αναφορά συγκεκριμένων ποσών. Γιατί αν ακυρώσουμε την ευελιξία, την ελαστικότητα, τότε τι κάνουμε. Γιατί όλοι ήρθαν με κάποια ιδέα σαφών ορίων και περιορισμών. Έτσι όμως θα μου πούν τα προηγούμενα μέσα, γιατί τα συγχωνεύσαμε. Οπότε θέλουμε να έχουμε περιθώριο ελιγμών, ευελιξία. Αυτό είναι σημαντικό, το που θέλουμε να το κρατήσουμε. Και στη συνέχεια θα περάσουμε στα άρθρα που δεν καλύπτονται από τη συμβαστική πρόταση. Αυτά, ευχαριστώ. Κύριο Σπαντσέρη, μία μόνο διευκρίνηση προς τον κύριο Γκάλερ, τον φίλο Γκάλερ. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε ουσιαστικά σε μια συμφωνία, σε μια ευρεία συμφωνία και για τα θέματα που αγύρισε, επί παραδείγμα, τη σχέση μεταξύ δημοκρατίας και ανθρωπινών δικαιώμα των... διευκρίνηση μόνο, αλλά είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το θερμόμετρο που μας δίνουν το μήνυμα εάν υπάρχει δημοκρατία σε ένα κράτος και τι τύπου, τι ποιότητας δημοκρατία. Γιατί μια δημοκρατία, ένα κράτος που έχει δημοκρατία σε τυπικού όρου, αλλά δεν σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα, δεν έχει δημοκρατία. Άρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μετρήσουμε, αλλά βέβαια και να συνδυάσουμε αυτό που λες και εσύ. Με αυτή τη διευκρίνηση όμως πολιτικής φύσεως οπωσδήποτε. Η κυρία Μακέβαν. Τελειώνει εδώ η συνεδρίαση. Ήταν μεγάλη μέρα. 4 Μαρτίου, 16 και 30. Έως 18 και 30 ψηφίζουμε τροπολογίες. Ευχαριστώ. Πέρα στη συνεδριάσεως.